εκφράζαμε την ανησυχία μας όσον αφορά τη δραματική κατάσταση στη Συρία. Λίγες ώρες μακριά από το Στρασβούργο οι Σύριοι υποφέρουν και είναι όμοιροι ενός παιχνιδιού που τους ξεπερνά. Οι πρόσφατες εξελίξεις τελευταίες ημέρες απομακρύνουν κάθε προοπτική ε, ειρήνευση. Σε λίγες εβδομάδες η επίθεση στην Ανατολική Γκούτα είχε ως αποτέλεσμα πάνω από χίλιους νεκρούς. Παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι, ευάλωτοι, ε, χιλιάδες τραυματίες βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης ανάγκης. Η κλιμάκωση της βίας αφήνει να σκεφτούμε τα χειρότερα. Η ανθρωπιστική κατάσταση στο εσωτερικό του θύλακα που είναι περικυκλωμένος μπορεί να επιδεινωθεί πολύ γρήγορα. Τα νέα που μας στάνουν από εκεί είναι φρικτά. Όλα τα μέρη οφείλουν να, να αναλάβουν τις ευθύνες τους συμπεριλαμβανομένου του ε, εγγυητή, των εγγυητών της διαδικασίας της ε, ε, ε, ΣΑΝΑ. Κανείς δεν μπορεί να δικαιολογήσει, τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βαρβαρότητα και τη σφαγή αθώων. Στο όνομά σας και στο όνομα του θεσμού μας θα κάνω μια επίσημη έκκληση για την εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Είναι επίγον για μια μόνιμη πάυση πυρός, είναι προσφύγων ώστε να προστατευτούν οι άοπλοι πολίτες. Επίσης, οι τραυματίες και οι άρρωστοι να μπορέσουν να, να εκενωθούν και να δρομολογηθεί βοήθεια. Είναι επίγον να βρεθεί μια πολιτική λύση μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γενέβης. Όλοι όσοι έχουν κάποια επιρροή θα πρέπει να δράσουν, να ενεργήσουν ώστε να πάψει αυτή η τραγωδία. Η ανθρωπότητα χάνεται στην Συρία. Ας μην χάσουμε και εμείς την ανθρωπιά μας. Πιστεύω πως αυτό το μήνυμα που φεύγει από το Στρασβούργο είναι ένα θετικό μήνυμα για τους πολίτες που βρίσκονται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 πιασμένοι στη μέση ανάμεσα στους ε, ε, μαχόμενους, είναι τα θύματα, είναι άοπλοι, δεν μπορούν να φύγουν από την πόλη. Ελπίζω πως χάρη σε αυτό το μήνυμα θα πιέσουμε προς σωστή κατεύθυνση. Και φέτος με την ευκαιρία της ημέρας των δικαιωμάτων της γυναίκας θα ήθελα να επιβεβαιώσω τη δέσμευση του Κοινοβουλίου στον αγώνα για την εξασφάλιση της πραγματικής ισότητας των δικαιωμάτων ανάμεσα στις γυναίκες και στους άνδρες. Και αυτό είναι ο του έτους, αλλά ακόμα πόρο απέχουμε από την νίκη. Τα στοιχεία μιλούν σαφώς, η, αδικία, η ανισότητα ε, εξακολουθεί να ισχύει και η παρουσία των γυναικών σε θέσεις ευθύνη είναι ακόμα ε, λιγοστή και φαίνεται να υπάρχει έλλειψη ακόμα σε φοιτήτριε σε τεχνολογικές και επιστημονικές σπουδές. Όπως επίσης δεν υπάρχει ισότητα ούτε μέσα στις οικογένειες. Σήμερα μόνο το 24% των μάνατζερ είναι γυναίκες και μόλις το 4,6% των διοικητικών σε υψηλά ιστάμενες θέσεις. Ε, Επίσης, 6,5 εκατομμύρια γυναίκες λιγότερες απασχολούνται από ότι άνδρες. Πιστεύω πως η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης, αλλά είναι και προς το συμφέρον της κοινωνίας μας. Στον κόσμο της εργασίας, οι γυναίκες αποτελούν ένα πολύτιμο πόρο. Έχει υπολογιστεί ότι αν αποκλειστούν οι γυναίκες από τον πραγματικό κόσμο, θα κοστίσει σε παγκόσμιο επίπεδο 11,5-3 μέχρι το 2025. Αυτό αντιστοιχεί στο ΑΕΠ της Ιαπωνίας, της Γερμανίας και της, ε, του Μεγάλου Βασιλείου. Ε, είναι σημαντικό να υπάρχει ισότητα ξεκινώντας από το μισθό για να εγγυηθούμε την ανάπτυξη και την απασχόληση σε ολόκληρη την οικονομία. Για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης χρειαζόμαστε γυναίκες επιχειρηματίες, επαγγελματίες, ε, πρωτοπόρες στην έρευνα. Αλλαγή νοοτροπίας είναι απαραίτητη, είναι ωστόσο αργή. Αλλά έχει ήδη ξεκινήσει. Το τελευταίο χρόνο έχει αυτοφανεί και μέσα από τον αγώνα κατά των στερεοτύπων για τον ρόλο των γυναικών όπως φαίνεται και από την εκστρατεία μη του. Ευχαριστώ τις συναδέλφους ε, Ρένκερ, Σλάιν και Μαρτέ που διοργάνωσαν ένα, ψηφίσμα, ένα μέσο από το οποίο συγκέντρωσαν υπογραφές που μου δόθηκαν ε, απόψε. Οι υπάλληλοι, οι άνδρες και οι γυναίκες που εργάζονται εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν συντάξει δικό τους, δική τους αναφορά με πάνω από χίλιες ε, υπογραφές και έλαβα το κείμενο αυτή της αναφοράς. Σας ενημερώνω ότι απόψε το γραφείο του, της Προεδρίας θα υιοθετήσει μια σειρά μέτρων για να προληφθούν οι σεξουαλικές παρανοχλήσεις εντός ε, του δεσμού μας. Ευχαριστώ και την Επιτροπή Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πολύτιμη και ακούραστη εργασία της υπέρ των γυναικών, όπως χαιρετίζω και το Ευρωπαϊκό Βραβείο για τις Γυναίκες στην ICT, το οποίο θέσπισε η Επίτροπος Γκάμπριελ και είναι ένα, απόδειγμα, ένα παράδειγμα Προς μίμηση. Η Ένωση θα πρέπει να αγωνιστεί για την πραγματική ισότητα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες γιατί δεν θα έχουμε καλύτερο κόσμο χωρίς να δώσουμε τη σωστή αξία στο ρόλο των γυναικών, στη δέσμευσή τους και το πάθος τους δεν πρόκειται για μάχη των γυναικών για τις γυναίκες ή κατά των ανδρών, αλλά πρέπει από κοινού άνδρες και γυναίκες να αγωνιστούμε γι' αυτό καθημερινά. Πολλοί δρόμος ακόμα πρέπει να διενηθεί, αλλά όλοι μπορούμε να παίξουμε το δικό μας ρόλο. Αυτό είναι νομίζω το καλύτερο μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τους πολίτες ε, επί τη ευκαιρία της 8ης Μαρτίου. Άρχεται η συνεδρίαση. Ο κύριος Μαριάς ζήτησε το λόγο, νομίζω. Κύριε Πρόεδρε, επί 12 ημέρες συνεχίζεται η παράνομη κράτηση δύο Ελλήνων στρατιωτικών στις φυλακές υψής της ασφαλείας της Αδριανούπολης στην Τουρκία. Είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινή γνώμη. Χθες σε ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο στην ορεστιάδα οι γονείς των δύο παλικαριών και οι κάτοικοι ζήτησαν την άμεση απελευθέρωσή τους. κάνω έκκληση στο σώμα και σε εσά προσωπικά όλοι μαζί με μια φωνή εδώ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να απαιτήσουμε από τις τουρκικές αρχές την άμεση απελευθέρωση των δύο ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται παράνομα στις τουρκικές φυλακές υψής της ασφαλείας της Αδριανούπολης. Θέλουμε την άμεση συμπαράστασή σας κύριε Πρόεδρε. Το αναμένει όλη η κοινή γνώμη. Το αναμένουν οι γονείς των παλικαριών. Ευχαριστώ. Προσωπικά θα παρακολουθήσω τι γίνεται και θα ζητήσω τα νεότερα από τον Τούρκο πρέσβη, ο, ο κύριος Γκόλνης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλήσατε για την ισότητα ανδρών και γυναικών και κατά της παρενόχλησης σεξουαλικής. Επειδή όμως μιλήσατε και για τους ε, δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλω να υπενθυμίσω κάτι που με ανησυχεί ιδιαίτερα. Μια Γαλλίδα υπάλληλο, η οποία εργάζεται στη Γενική Γραμματεία, είχε ξεκινήσει με κατηγορίες, πάρα πολύ σοβαρές κατηγορίες, οι οποίες ίσως να είναι και αβάσιμες, δεν αμφισβητώ αυτό, κατά ενός υψηλόβαθμου υπαλλήλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον οποίο δεν θα κατονομάσω. Το μήνυμα που έστειλε έχει σβηστεί από την διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο, καθότι αυτό έγινε στα προσωπικά μας ε, ε, ηλεκτρονικά μηνύματα. Εάν οι κατηγορίες αυτής της γαλίδας υπαλλήλου είναι αβάσιμες, φυσικά και ο υψηλόβαθμος αυτός υπάλληλος ο οποίος κατηγορείται πρέπει να απαντήσει ή πρέπει να δοθεί μια απάντηση επίσημη από μέρους του Προέδρου αυτού του Κοινοβουλίου. Όποια και να είναι όμως η ουσία αυτής της υπόθεσης, θεωρώ ότι είναι εντελώς απαράδεκτο να υπάρχει παρέμβαση στους προσωπικούς υπολογιστές όλων των μελών αυτού του Κοινοβουλίου για να σβηστεί αυτό το μήνυμα αυτής της υπαλλήλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Γκόλνης. Θα το επαληθεύσουμε αυτό που μου είπατε. Σας Θα μας δώσετε όλα τα τεκμήρια που έχετε στη διάθεσή σας και μετά θα δούμε. Ο κύριος Μιράντα παρακαλώ. Η κυρία Μιράντα. Κύριε Ταγιάννη, ζητώ το Κοινοβούλιο μας επί τη βάση του άρθρου 7 του κανονισμού να στραφεί προς τις Ισπανικές Αρχές και να εκφράσει την ανησυχία του για την κατάσταση του κυρίου Ουριόλ Χουνκέρας Βές που είναι πολιτικός κρατούμενος αυτή τη στιγμή. Ναι. Ο κύριος Γιούρικ. Κύριε Πρόεδρε, μια μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου απευθύνθηκε στον προκάτοχό σας, τον κύριο Σούλτς και εκατόπιν σε εσάς σε σχέση με έναν πίνακα ζωγραφικής που εκτίθεται σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο, έναν όροφο πιο κάτω, με τον προκλητικό τίτλο «Ντολορόζα». Πρόκειται για προσβολή της πίστης ε, πολλών εξημών, αλλά περιέχονται και ιερά σύμβολα από την παράδοση της Ευρώπης. Της Ευρώπης. Πρόκειται για μια ταπείνωση, το είπαμε ξεκάθαρα, αλλά προφανώς εσείς συμφωνείτε με αυτό. Αλλά εδώ πέρα προσβάλλεται και η Παναγία. Είναι μεγάλη σαρακοστή και είναι νομίζω μια ευκαιρία για σας να τερματίσετε αυτήν την κατάσταση. Απευθύνω έκκληση στην τιμή σας, όπως έκανα και στον προκατοχό σας. Θα ασχοληθούμε με αυτό, με το αρμόδιο όργανο, ο κύριος Τουργάις. Σας ευχαριστώ κύριε Ταγιάννη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που θυμίζετε. Ε, θέλω να θυμίσω στην κυρία Μιράντα ότι στην Ισπανία δεν υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι. Υπάρχουν ε, ε οι εγκληματίε, οι εγκληματίε που έκαναν πραξικόπημα. Αν θέλετε να. Ναι, ναι, αυτό είναι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι και δεν είναι πολιτικοί κρατούμενοι, δεν υπάρχουν σε μια δημοκρατία όπως η Ισπανική Δημοκρατία. Προχωράμε στην ε, ημερήσια μαζί